Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίασή μα είναι διαθέσιμα πλέον. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε παρατηρήσει ε, επ' αυτών. Όχι από ό,τι βλέπω. Άρα εγκρίνουν τα πρακτικά και περνάμε στην ψηφοφορία. Και